Σας ευχαριστώ για την ε, υπομονή σας και μετά το διάλειμμα επανερχόμαστε. Έχουμε και τον καλεσμένο μας, τον κύριο Εμμανουέλ, ο οποίος θα παρουσιάσει τη συνέχεια την ε, συνέχεια της ε, αξιολόγησης του βαθμολογίου για τα θέματα δικαιοσύνης Θυμόσαστε ότι το Μάρτιο είχε λάβει χώρα μια ανακοίνωση της Κομισιόν για το βαθμολόγιο της ε, δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί τη βάση του έργου της Επιτροπής για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ήταν αυτή που είχε προκαλέσει ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου η Κομισιόν όπου ζητήθηκε μάλλον από την Κομισιόν να διευρύνει το πλαίσιο του αθμολογίου για να καλύψει και την ποινική δικαιοσύνη και την αμοιβαία αναγνώριση και εμπιστοσύνη. Ο κ. Κράμπιτ λοιπόν έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις 17 Μαρτίου η Κομισιόν παρουσίασε <clears throat> τη δεύτερη έκδοση του αθμολογίου για τη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτό είναι ένα εργαλείο Πληροφόρηση δίνει μια συγκριτική επισκόπηση της λειτουργίας των εθνικών δικαιακών συστημάτων. Το βαθμολόγιο αυτό έχει σε στόχο να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να επιτύχουν πιο αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης με το να δώσει αντικειμενικές και, αντικειμενικά και αξιόπιστα στοιχεία για την ποιότητα, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος δικαιοσύνης έχει σαν στόχο να διαερευνήσει δυνητικές βελτιώσεις, να δει προβλήματα κτλ. Δεν είναι βέβαια ένα είδος καλυστίου μεταξύ των κρατών μελών, δεν συγκρίνει την ποιότητα μεταξύ κρατών μελών, αλλά έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει μια βελτίωση. Η Κομισιόν αποφάσισε να δημιουργήσει αυτό το εργαλείο για διάφορου λόγου. Καταρχήν, η αποτελεσματικότητα τη εθνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο είναι κέρδιο για την αποτελεσματικότητα τη εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε υπάρχει το δικαίωμα αποτελεσματικής θεραπείας ενώπιον δικαστηρίου που αναφέρεται στο άρθρο 14 της Χάρτας Ανθρωπή ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και είναι σημαντική επίσης και αυτή η αποτελεσματικότητα δικαιοσύνη για την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών και δικαστικών αρχών και η αποτελεσματικότητα επομένως είναι και ένας τρόπος για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική σταθερότητα. Τα εθνικά συστήματα λοιπόν απόδοση δικαιοσύνη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την εμπιστοσύνη και στην οικονομία και να εξασφαλίσουν την οικονομική ανάπτυξη. Από το 2012, για τον λόγο αυτό, η βελτίωση της ποιότητας και της ανεξαρτησίας καθώς και της αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης αποτελεί μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Κομισιόν αν, ανατέμνει τις διαφορετικές αλλαγές και όπου είναι απαραίτητο προτείνει συστάσεις για το απαιτούμενο σε σχέση με τη βελτίωση στους τομείς αυτούς. Το βαθμολόγιο δικαιοσύνης ε, συμβάλλει στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και στις αναλύσεις αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι μία ασθενής απόδοση στο βαθμολόγιο θα πρέπει να προκαλέσει και μία βαθύτερη ανάλυση των λόγων που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Πάντα υπάρχει και μία αξιολόγηση η οποία είναι ειδική αναχώρα, η οποία γίνεται με διμερείς διαλόγους με το εμπλεκόμενο κράτος μέλος και λαμβάνει υπόψη το, η λειτουργία του συστήματος στην χώρα αυτή, του νομικού συστήματος, όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες λαμβάνονται υπόψη. Το βαθμολόγιο λοιπόν είναι μονάχα ένα συνεκτιμούμενο στοιχείο το οποίο θα ληφθεί υπόψη για τα θέματα αυτά και η υποστέμενη του αξία είναι ότι δίνει ένα συγκριτικό μια συγκριτική επισκόπηση σε σχέση με τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Αυτές λοιπόν οι αξιολογήσεις που γίνονται επί τη βάση επί τη βάση του βαθμολογίου δικαιοσύνη μπορούν να οδηγήσουν την Κομισιόν να κάνει συγκεκριμένε για κάθε χώρα συστάσεις και το Συμβούλιο θα πρέπει στη συνέχεια να εγκρίνει αυτές τις ε, συστάσεις. Δέκα κρατημέλη το 2013 ε, είχαν να αντιμετωπίσουν ειδικέ συστάσεις που τους ενεθάρρυναν να βελτιώσουν το σύστημα απόδοσης δικαιοσύνης. Ποια είναι τώρα τα κύρια στοιχεία του βαθμολογίου του 2014, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με το θέμα της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της απόδοσης δικαιοσύνη. Όπως ξέρετε, τα τρία κέρια κεφάλαια του βαθμολογίου είναι αποτελεσματικότητα, ποιότητα και ανεξαρτησία του συστήματος δικαιοσύνης. Για το θέμα της αποτελεσματικότητας, το βαθμολόγιο εξετάζει το μήκος της διαδικασίας, τη διάρκεια τη διαδικασία. για ε, διοικητικές ή αστικές υποθέσεις, την ικανότητα των δικαστηρίων να αντιμετωπίσουν το φόρτο εργασίας, ακόμα και αυτά τα οποία προέρχονται από προηγούμενα έτη. Το συμπέρασμα είναι ότι ορισμένα κατημέρια εξακολουθούν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερε προκλήσει σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του συστήματο δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει μάκρο διαδικασία σε πρωτόδικο επίπεδο και χαμηλό ποσοστό ε, περάτωση των διαδικασιών και μεγάλο αριθμό εκκρεμών διαδικασιών. Το θετικό είναι ότι ο αριθμός των κρατών, πολλές κράτες, χώρες μέλη είναι σε φάση ε, εφαρμογής μεταρρυθμίσεων για το σύστημα δικαιοσύνης τους για να βελτιώσουν τη λειτουργία αυτού του ιδίου συστήματος. Το αποτέλεσμα όμως των ε, φιλοδόξων αυτών μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει σε πολλά κράτη-μέλη δεν μπορεί ακόμα να αξιολογηθεί γιατί το βαθμολόγιο του 2014 χρησιμοποιεί στοιχεία του 2012 και χρειάζεται χρόνος για μια μεταρρύθμιση στον χώρο της δικαιοσύνης και χρειάζεται χρόνος για να δούμε θετικά αποτελέσματα. Αλλά έχει ετήσιο χαρακτήρα το βαθμολόγιο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι τα θετικά αποτελέσματα της μεταρρύθμισης θα μπορούν να γίνουν πιο ορατά μέσω του βαθμολογίου για το θέμα της ποιότητας του συστήματος δικαιοσύνης στο βαθμολόγιο χρησιμοποιεί ορισμένους ενδείκτες ροής που είναι παράμετροι που συμβάλλουν στην ποιότητα του συστήματος δικαιοσύνης. Παραδείγματος χάρη εκπαίδευση των δικαστικών που είναι πολύ σημαντική και επίσης η χρήση πληροφορικής και τεχνολογιών αυτού του είδους και τη σχέση μεταξύ διαδίκων και δικαστηρίου. Επίσης πληροφορίες σε σχέση με την ε, ε την αποτελεσματικότητα της διαιτησίας. Σας υπενθυμίζω ότι ένα πρόσφατο ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για εξοδικαστικές επιλύσεις ε, αντιδικιών 80% από αυτούς που απάντησαν στο Ευρωβαρόμετρο είπαν ότι θα θέλανε μια εξωδιαδικαστική συμβαστική λύση και μόνο 8 είπαν θα πάνε ούτως ή άλλως στο δικαστήριο. Υπάρχουν και στοιχεία για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους. Το τελευταίο στοιχείο είναι η ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών για πρώτη φορά το βαθμολόγιο ξεπερνάει την απλώς παρουσίαση των αντιλήψεων σε σχέση με αυτή την ανεξαρτησία του Εθνικού Συστήματος Δικαιοσύνης και τα γραφήματα αυτά παρουσιάζονται επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα του περσινού βαθμολογίου ότι δηλαδή υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε σχέση με την ε, αντίληψη ανεξαρτησίας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης. Για να ξεπεράσουμε όμως μονάχα το θέμα των αντιλήψεων, το βαθμολόγιο του 2014 παρουσιάζει την ε, Ε, κατάσταση του νομικού πλαισίου που έχει σε στόχο την εξασφάλιση της δικαιοσύνης. Στο μέλλον θα θέλαμε μαζί με το δίκτυο των δικαστικών αρχών, δικαστικών και εισαγγελέων και μαζί με τα κράτη-μέλη θα θέλαμε να καθορίσουμε πώς μπορεί το βαθμολόγιο αυτό να εξετάζει τα συγκριτικά στοιχεία και να δημιουργήσει συγκριτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του δικαστικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Ο πίνακα αποτελεσμάτων το 2014 λαμβάνει υπόψη το ποια χώρα αξιολογήθηκε στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2014 και ένα από τα συμπεράσματα του προσπατότερου πίνακα είναι ότι και πάλι υπάρχει ε, κενό στην ε, υποβολή πληροφοριών. Πρέπει λοιπόν όλοι να φροντίσουν να δίνουν περισσότερα στοιχεία για τα θέματα αυτά. Όπως θα δείτε και στον πίνακα αποτελεσμάτων από τις γραφικές παραστάσεις, δεν υπήρξε δυνατότητα συλλογής κάποιων στοιχείων για αρκετά κράτη-μέλη. Έγινε λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια για να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτό το κενό, αυτή την έλλειψη των πληροφοριών. Ω προ αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εντείνει τι προσπάθειέ τη σε συνεργασία με τα τις ομάδες επαφής που δημιουργήθηκαν το 2013. Η ομάδα των προσώπων επαφής από τα κράτη-μέλη εκπροσωπεί όχι μόνο τα Υπουργεία Δικαιοσύνη αλλά και το δικαστικό κλάδο. Επικεφαλής ε, της ομάδας αυτής μας λένε ότι μπορεί να βρεθεί λύση στην ε, υποβολή, στην καλύτερη υποβολή συγκρίσιμων δεδομένων. Και όπως είπα, ως προς την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα ζητήματα αυτά. Ε, εν είδη συμπεράσματος, Πρόεδρε, όπως είπατε, να ευχαριστήσω και πάλι το Ευρωκοινοβούλιο και την Επιτροπή σας και όλες διατηρήσει την κυρία για την πολύ θετική σας τάση και τη θετική έκθεση που δημοσιεύτηκε. Αλλά και το σχετικό ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα σε ό,τι αφορά τον πίνακα αποτελεσμάτων ε, για, την Ευρωπαϊκή, για τη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό για μας και είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βλέπει ότι το Ευρωκοινοβούλιο θέλει να προχωρήσει. Θέλει να αναπτύξει περαιτέρω τον ε, πίνακα αποτελεσμάτων για τη δικαιοσύνη. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτού του είδου τη θετική ενέργεια για ένα ζήτημα που ενδιαφέρει όλου μα από κοινού για την λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για τη στήριξή σας. Και σας διαβεβαιώνω ότι θα επιδιώξουμε να βελτιώσουμε τον πίνακα αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ήταν πραγματικά μια πολύ καλή αποτίμηση του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου, ιδίως του ρόλου της Επιτροπής μας και σωστά επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση του πίνακα αποτελεσμάτων ε, έπρεπε να έχει περιληφθεί στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν και καλώς περιληφθεί. στην τελική φάση της θητείας. Και στο τέλος εφαρμογής του προγράμματος της Στοκχόλμης θα γνωρίζετε ότι και αυτό δεν ήταν απλό. Διότι υπήρξε διαφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων, <clears throat> πέραν τη συζήτηση για τα διάφορα συστατικά τμήματα του συγκεκριμένου ε, θέματος. Ήταν λοιπόν μεγάλη σημασία, ιδίω για την Επιτροπή Ελευθερίων του Πολίτη. Και τώρα, χρόνος για συζήτηση. Κυρία Γκόντς, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την έκθεση. Θα ήθελα να παρατρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της. Ήταν ε, πραγματικά πολύ θετική ιδέα να εισαχθεί ο πίνακα αποτελεσματών για τη δικαιοσύνη μαζί με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και παρά το πακέτο της έκθεσης πρέπει να πω ότι εκτιμώ ιδιαιτέρως τη διάρθρωση της συνιστώσας για την ε, ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα είπατε κι εσείς ότι μελετήσατε και το πώς γίνεται αντιληπτή η ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου. Είναι σημαντική η εξέλιξη αυτή και να πω ότι στην έκθεσή μου που είχε ευρεία στήριξη και εγκρίθηκε με ισχυρότατη πλειοψηφία στην Ολομέλεια να πω ότι εκεί απευθύνεται έτοιμα να πάμε ακόμη περισσότερο, ακόμη πιο μακριά και να συμπεριληφθεί και το σύστημα ποινική δικαιοσύνη των ε, πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε επανειλημμένως συζητήσεις, καθώς προετοιμάζαμε την έκθεση αυτή, για το πόσο είναι απειλή η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου. Και είπαμε ότι το πρόβλημα δεν είναι εδώ η απλοποίηση του ποινικού δικαίου, η ευθυγράμμιση του, αλλά οι διαδικασίες. Άλλα ζητήματα επίσης, όπως η διαφθορά, στην έκθεση αυτή τονίζεται η σημασία τους. Πρέπει να συμπεριληφθεί όντω και το ποινικό δίκαιο στον πίνακα αποτελεσμάτων. Ε, ένα άλλο θέμα στην έκθεση αυτή είναι οι μηχανισμοί ε, επιβολής του νόμου για μια εύστοχη αποτίμηση αλλά και τους μηχανισμούς που εφαρμάζονται. Ξέρω ότι στις σχετικές ανακοινώσεις οι μηχανισμοί αυτοί περιγράφονται επαρκώς. Επίσης στην έκθεση αυτή καλώς λέγεται ότι θα ήταν καλό να υπάρχει διαχωρισμός των δύο κάποια στιγμή. Ένας μηχανισμός επιβολής του νόμου από τη μια και ένας πίνακας αποτελεσμάτων της δικαιοσύνης από την άλλη. Νομίζω λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για τις επιμέρους χώρες ε, να έχουν αυτές τις επιμέρους αναχώρα τάσης. Κανεί δεν αρέσει, δεν θέλει βέβαια να παραδέχεται τι αδυναμίε του, όμω είναι ένα μέρο του συστήματο πολύ απαραίτητο και πρέπει να περιλαμβάνεται όπω σωστά έγινε. Το επισημαίνει και η έκθεσή μα. Ευχαριστώ πολύ. Άλλα σχόλια, κύριε Μπρόγκ. Η προσέγγιση του πινάκα αποτελεσμάτων δίνει μια μεγάλη δώσει αντικειμενικότητας στην όλη διαδικασία. Όμως, ίσως να υπάρχουν ε, ελλείψεις ε, ή μειονεκτήματα στο νομικό σύστημα που δεν βρίσκουν την ε, απήχησή του στον πίνακα αποτελεσμάτων. Λόγω χάρη δεν θα μπορούσε κανείς να αναρτηθεί για το πόσοι πολιτικοί ασκούν προεκλογική εκστρατεία στις διάφορες χώρες και έχουν υποστεί και κάποια δίωξη πόσοι πολιτικοί επίση της αντιπολίτευσης ε, βρίσκονται στη φυλακή με εκκρεμωδικία και χωρί να πλησιάζει η ημερομηνία εκδίκαση τη υποθεσή τους. Αυτά τα βρίσκω πολύ σημαντικά στοιχεία, διότι όταν οι κυβερνήσεις κάνουν κατάχρηση της εξουσία τους, συνήθως την κατάχρηση την κάνουν κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Αυτό καλό θα ήταν να πηχείται και στον πίνακα αποτελεσμάτων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Άλλα σχόλια. Άλλα σχόλια για τον πίνακα αποτελεσμάτων. Όχι. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Γκράμπιτ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ κυρία Γκόντς ε, για την υποστήριξή σας. Πράγματι, η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος είναι ένας τομέας όπου πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Είναι ένα θέμα περίπλοκο και πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια του δικαστικού σώματος όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι ενδιαφερόμενοι θα σημειώσουν πρόοδο. Η ποινική δικαιοσύνη. Είναι δεδομένου ότι ο στόχος αυτού του πίνακα των αποτελεσμάτων είναι να βοηθήσει και εκείνο το οποίο ε, ε, αποσκοπεί είναι ε, να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλους τους τομείς. Είναι όμως ένα μέσο που εξελίσσεται και πρέπει να δούμε πώς μπορεί να επεκταθεί αυτός ο πίνακας αποτελεσμάτων στο τομέα τη δικαιοσύνη σε, σε όλους τους τομείς. Στο τέλος του 2014, του 2013 με συγχωρείτε, εξηγήσαμε ότι θα εξηγήσουμε πώς θα συλλέξουμε στοιχεία από τους πιο κρίσιμους τομείς κυρίως για τα εγκλήματα, τα οικονομικά εγκλήματα. Εδώ υπάρχει σχέση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε, δηλαδή ότι υπάρχει δυνατότητα να διευρύνουμε τον τομέα αυτό, αλλά εάν δείτε πόσο δύσκολο είναι να αποκτήσουμε στοιχεία από απλές ποινικέ διαδικασίες, ακόμα και στον αστικό και εμπορικό τομέα, να έχουμε δείκτε σε αυτούς του τομεί, είναι πολύ πιο δύσκολο να αποκτήσει κανείς δείκτε για 28 κράτη-μέλη. Και αυτή είναι μια πρόκληση, δηλαδή θα πρέπει να συλλέξουμε στοιχεία για τα 28 κράτη-μέλη. Η προστιθέμενη αξία αυτού του πίνακα είναι ότι έχει μια, ένα, ένα συγκριτικό πίνακα και πρέπει να το δούμε με ρεαλιστικό τρόπο ε, βλέποντας ποια είναι η διαθεσιμότητα στοιχείων στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερε δυσκολίες, τι μεγαλύτερε προκλήσεις σε αυτό το τομέα. Τώρα, για το θέμα που έδειξε ο κ. Μπρόγκ, νομίζω ότι αυτό έχει περισσότερη σχέση με το ποινικό δίκαιο και όχι με το ευρωπαϊκό εξάμεινο και δεν νομίζω πρέπει να σας πω, δεν νομίζω να έχετε αμφιβολία ότι εδώ είναι πολύ δύσκολο να βρούμε συγκριτικά στοιχεία. Σε αυτό το τομέα, πάντοτε για 28 κράτη-μέλη. Αυτή είναι μια πραγματική δυσκολία για όλους μας και θα πρέπει να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την ικανότητα συλλογής δεδομένων και συνεργαζόμαστε ε, με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΠΕΖ και γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια μεγάλη δυσκολία. Στο παρόν στάδιο προσπαθούμε να παγιώσουμε την εμπειρία μας ε, στην ποινική, διοικητική και εμπορική δικαιοσύνη και βλέπουμε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας, αλλά πάντοτε ε, υπό την προπόθεση θα έχουμε σωστά στοιχεία και θα μας παρέχονται νέες πληροφορίες. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Πολύ καλά. Νομίζω ότι τελειώσαμε και με αυτό το θέμα της εμερικής διάταξης. Προχωράμε τώρα στην κοινή συζήτηση σημεία 12 και 13 όσον αφορά ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις συνθήκες κράτησης της φυλακές στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αντιπροσωπεία Λίμπε στην Ιταλία σχετικά με την κατάσταση στις φυλακές και στα σοφρονιστικά ιδρύματα. 26-28 Μαρτίου 2014 έγινε αυτή η επίσκεψη. Είχαμε την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης, το οποίο εγώ συνέταξα ως πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και ως επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας που πήγε στην Ιταλία. Από τις 26-28 Μαρτίου φέτος εγώ ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, στην Ιταλία για την κατάσταση που επικρατεί στι φυλακές και τα σοφρονιστικά ιδρύματα. Όπως σα είπα, ήμουν πρόεδρος αυτής τη Επιτροπής, ήταν η κυρία Γκάντ, ο κύριος Έγγελ και ο κύριος Γιακολίνο ω ε, συνοδός ο σκοπός αυτής της αντιπροσωπεία ήταν να αξιολογήσει την κατάσταση στις, οφρονιστικές στις φυλακές και στα σοφρονιστικά ιδρύματα της Ιταλίας και να αξιολογήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων μας την πρόοδο που έχει επιτελεστεί από την Ιταλία για να συμμορφωθεί με ε, την απόφαση ρετζιάνι, την πιλωτική απόφαση Ρετζιάνι ε, στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Ήταν αυτή η απόφαση το Ρεγκιάνι, την οποία γνωρίζετε ίσως, η οποία δήλωσε, σύμφωνα με αυτή την απόφαση, δηλώθηκε ότι οι συνθήκες στις φυλακές στην Ιταλία δεν ήταν σύμφωνες με το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αναφέρεται στην απαγόρευση ε, των βασανιστήριων και απάνθρωπη μεταχείριση των κρατουμένων. Το γεγονός ότι είναι ασφικτική κατάσταση φυλακές ε, δεν μπορούν οι κρατούμενοι να ζουν υπό ανθρώπινες συνθήκες. Γι' αυτό αποφάσισε η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, οι συντονιστές της συγκεκριμένα, να υποβάλουν μια έκθεση και να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές στα κράτη-μέλη. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνη η Ιταλία όσον αφορά τις κακές συνθήκες φυλάκισης. Σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντοτε, υπάρχουν προβλήματα ε, ως προς τις εγκαταστάσεις στις φυλακές και οι συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων είναι προβληματικές διότι υπάρχει υπερπληθυσμός στις φυλακές και αυτό είναι ένα πρόβλημα σε πολλά κρατημέλη. Δεν είναι λοιπόν μόνη η Ιταλία σε αυτό το πρόβλημα, δεν θεωρείται ως μεμονωμένη εμπειρία, αλλά υπάρχουν παράλληλα παραδείγματα αυτής της δυσάρεστης κατάστασης και των προβλημάτων που πρέπει να συζητήσουμε, εάν θέλουμε, να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας ως μέλη της Σύμβασης των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε σωστά τους φυλακισμένους. Λοιπόν, ε, όταν ε, ψηφιστεί το επόμενο κοινοβούλιο μπορεί να υπάρξουν και άλλες ε, επισκέψεις ε, φυλακές άλλων κρατών μελών και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία με την Επιτροπή για να αποτρέπονται τα βασανιστήρια και να συνεργαστούμε με άλλα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σήμερα υπάρχει ο ειδικό σύμβουλος του Ιταλού Υπουργού Δικαιοσύνη και πρόεδρος τη ειδική Επιτροπής για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των φυλακών. Είναι εδώ ο κύριος Μάρο Πάλμα. Θα τον ακούσουμε και έχετε το σχέδιο έκθεσης το οποίο κυκλοφόρησε που έστειλε το γραφείο μου και η Επιτροπή ε, Λίμπε. που δικαιολογεί την επίσκεψη της αντιπροσωπείας στην Ιταλία και την απόφαση του Ρεγκάνη. Ε, όλοι οι νομικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Υπάρχει το πιάνο κάτσερι, δηλαδή υπάρχει ένα σχέδιο φυλακών στην Ιταλία. Το πρώτο σύνολο μέτρων που υιοθετήθηκαν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή την δυσάρεστη κατάσταση στις ορισμένες τελικές φυλακές, να περιοριστεί ο αριθμό των κρατουμένων, να εισαχθεί ένα σύστημα ε, προληπτικών και διορθωτικών μέτρων, ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με την ομοθεσία για τα ναρκωτικά και όσον αφορά την επιβολή βασανιστήριων στις φυλακές και άλλα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά με την αμνηστία, την, ε, την απονομή χάριτος. προκειμένου να γίνει γνωστή η κατάσταση την οποία εμείς ζήσαμε με προσωπικά μετά από την επίσκεψη στη φυλακή Ραμπίμπια στη Ρώμη, Κάτζα σε κόντα Φεμιλίδα, είναι γυναικείς φυλακές, Ραμπίμπια, καθώς και τη φυλακή Ποντζορεάλε στην Νάπολη. Υπάρχουν ορισμένα συμπεράσματα τα οποία, στα οποία καταλήξαμε και θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας συνοψίζοντας. Το είπα δημόσια άλλωστε εντυπωσιάστηκα, συγκινήθηκα βαθιά και εξεπλάγιν τρόμαξα από τις συνθήκες αυτή τη φυλακή Πότζο Ρεάλε. Πρέπει να πω ότι ήταν φρικιαστικές, πραγματικά. Το είπα και στην Υπουργό Δικαιοσύνη. Έχω δει πολλές φυλακές στη χώρα μου, αλλά όχι μόνο στη χώρα μου. Ποτέ όμως δεν είδα κάτι τέτοιο όπως το Πόρτο Ρεάλε. Ποτέ. Ε, για την απόφαση του Ρετζιάννη ε, η βάση ήταν ότι δεν μπορεί να κρατάει κανείς εννέα άτομα 22 ώρες την ημέρα τουλάχιστον μέσα σε ένα χώρο 10-12 τετραγωνικών. 9 άτομα μαζί να κρατούνται σε ένα τόσο μικρό χώρο. Σε ένα χώρο, σε ένα κελί 12 τετραγωνικών. εννεα άτομα ενα χωρο σε ενα κελι 12 τετραγωνικων εννεα ατομα μαζι τα οποία ζουν, κοιμούνται, τρώνε μαζί 22 ώρες την ημέρα, χωρίς ε, δυνατότητα άθλησης, ε, χωρίς ε, τίποτα να τους προσφέρεται, από πλευρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή επαγγελματικής κατάρτισης. Ήταν μια εντυπωσιακή σκηνή αυτή που είδαμε εκεί. Γι' αυτό δεν απορίες άξιο το γεγονός ότι αυτές οι συνθήκες θεωρήθηκαν ως βασανιστήρια. Έτσι αποφάσισε ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η κατάσταση ήταν τρομακτική. Εκτιμούμε όμως τις προσπάθειες που καταβάλει η Ιταλική κυβέρνηση προκειμένου να επιφέρει βελτιώσεις στις φυλακές αυτές ιδέες που διατυπώθηκαν και θα πρέπει να υλοποιηθούν, όπως ε, σχετικά με τους κρατουμένους, μια εγγύηση θα πρέπει να υπάρχει για καλές συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων και θα υπάρξει να υπάρχει ο υπερασπιστής των δικαιωμάτων των κρατουμένων, ένα είδος ε, συνηγόρου όπως ο συνήγορος του πολίτη δεν είναι ο συνήγορος του κρατουμένου και ολοκληρώσαμε την έκθεσή μας καταδικάζοντας οποιαδήποτε πράξη βίας μέσα στο χώρο των φυλακών και παροτρύνουμε την Ιταλική κυβέρνηση να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα που οφείλονται στον υπερπληθυσμό των κρατουμένων. Είναι μια κατάσταση συστημική στην Ιταλία αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, τώρα κυκλοφόρησε αυτό το έγγραφο όπως είπαμε, είναι στη διάθεσή σας. Θα μας μιλήσει ο κ. Μαύρο Πάλμα και κατόπιν ίσως μπορούμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Ο Πάλμα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με καλέσατε και πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω πολλαπλώς και την Επιτροπή σας για την ε, επίσκεψη που κάνετε στις Ιταλικές φυλακές. Είναι μια νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής σας στην παρακολούθηση της κατάστασης τους χώρους στέρησης της ελευθερίας στην Ευρώπη. Για μένα αυτό είναι μια πολύ καλή και θετική εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Επιτροπής σας και <clears throat> ελπίζω όπως αναφέρετε και στις συνιστάτε στην έκθεσή σας να διευρυνθεί και να συνεχίσει αυτή η δραστηριότητα και από το νέο κοινοβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές. Όπως είπατε προηγουμένως, η Ιταλία αντιμετωπίζει μια πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί το σοφρονιστικό της σύστημα όπως ε, αναφέρεται στην έκθεση, δεν συνάδει με μία από τις πιο βασικές υποχρεώσεις στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, που είναι το άρθρο 3 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Υπάρχει λοιπόν μία απόλυτη υποχρέωση ότι θα πρέπει να, θα πρέπει να αποτρέπονται πλήρως οι κακομεταχειρήσεις και οι βασανισμοί για να σας πετιμήσω τις προηγούμενες δραστηριότητες μου για πάρα πολύ καιρό ήμουνα επικεφαλής Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστήριων και επομένως το έργο μου ήταν η παρακολούθηση των συνδικών κράτησης σε όλη την Ευρώπη για να, για να διακριβώσω κατά πόσο τα κράτη-μέλη τηρούσαν τις υποχρεώσεις σας, τις υποχρεώσεις τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι για μένα στην ε, θέση που βρίσκομαι και εκπροσωπώ την Ιταλική κυβέρνηση να προσπαθήσω <clears throat> να τροποποιήσω το σύστημα φυλακών στην Ιταλία από μια ε, κατάσταση που έχει παραβιάσει, που θεωρείται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις τους. Η δική μου λοιπόν θέση είναι τέτοια ώστε θεωρώ πρέπει να λάβουμε υπόψη το, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως μια ευκαιρία να αλλάξουμε το υπόδειγμα που επικρατεί στο Ιταλικό σοφανιστικό σύστημα και να περάσουμε από ένα σύστημα όπου η κράτηση είναι το κύριο σημείο εστίασης σε ένα σύστημα όπου αυτό το οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η επανενσωμάτωση των κρατουμένων στην κοινωνία. Είναι πολύ δύσκολο να περάσουμε από ένα σύστημα που βασίζεται στην αυστηρή στέρηση ελευθερία σε ένα σύστημα το οποίο εστιάζει την προσοχή του στην επανενσωμάτωση των κρατουμένων στην κοινωνία. Οι ενέργειες λοιπόν που έχουμε θέσει σε κίνηση σε αυτή τη διαδικασία είναι τέσσερις. Πρώτα απ' όλα, να μειώσουμε τον αριθμό των ατόμων που είναι σε κράτηση στις φυλακές με το να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε εναλλακτικές μορφές έκτησης ποινή να, με το να μειώνουμε την καταφυγή σε φυλάκιση και προφυλάκιση και με το να μην θεωρούμε τη θέση της ελευθερίας ως την μοναδική κύρωση που προβλέπεται από το ποινικό μας σύστημα. Η πρώτη μας λοιπόν πρόκληση είναι να μειώσουμε τον αριθμό των κρατουμένων. Από 69.000 έχουμε κατέβει σε 60.000 κρατουμένους τα τελευταία χρόνια. Η δεύτερη πρόκληση όμως είναι ακόμα πιο σημαντική. Αυτό είναι μια αλλαγή στο υπόδειγμα κράτησης. Αυτό που είδατε λοιπόν στο Πότζο Ρεάλε είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει ποτέ να μπορεί να λαμβάνει χώρα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα έπρεπε να ανήκει στο παρελθόν για οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αν οι κρατούμενοι σε μια φυλακή όπως το Πότζο Ρεάλε ήταν λίγοι, αν ήταν μικρός ο πληθυσμός των φυλακών, ακόμα και αν είχαν πάνω από 3-4 τετραγωνικά μέτρα ο καθένας τους, το πρόβλημα είναι ότι εξακολουθούν για ένα υπερβολικό αριθμό ωρών, 20-22 ορών να είναι έγκλειστοι και αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται δεκτό σε καμία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό φυσικά συμπεριλαμβάνει την Ιταλία. Η δεύτερη πρόκληση λοιπόν για μας είναι πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το μοντέλο που ακολουθούν τα σοφρονιστικά ιδρύματα και να τηρήσουμε απόλυτα τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις φυλακές. Το τρίτο θέμα είναι το κατά το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερους κρατούμενους σε πιο ανθρώπινες συνθήκες από διαρθωτική άποψη. Πολλές φυλακές είναι επεπαλαιωμένες, θα πρέπει να ανακαινιστούν, θα πρέπει να ανακατασκευαστούν για να δίνουν πιο πολύ προσωπικό χώρο διαβίωσης και όχι μονάχα ε, περισσότερα κελιά για τους κρατουμένους. Και το τέταρτο θέμα είναι η εισαγωγή ενός διπλού συστήματος θεραπείας. Μία ε, προληπτική θεραπεία και μία αντισταθμιστική θεραπεία. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΕΔΑΤ και ακολουθούμε αυτό το δρόμο. Μπορώ να δω ήδη κάποια αποτελέσματα. Ανέφερα στην αρχή ότι μειώθηκε ο αριθμός των κρατουμένων. Βλέπω να υπάρχει ένα νέο σύστημα εθνικών θεραπείων όταν πρόκειται για παραβίαση κάποιο από τα θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων. Ελπίζω δε ότι συντόμως η κυβέρνηση της Ιταλίας θα παρουσιάσει ένα διάταγμα για αυτούς οι οποίοι εκτείουν ποινές που, που σε σχετίζονται με αδικήματα που έχουν να κάνουν με τα ναρκωτικά, κατοχή ή εμπορία ναρκωτικών για να λάβει υπόψη και την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου που θεώρησε αντισυνταγματικό το νόμο σε σχέση με τις ποινές που επιβάλλονται σε αδικήματα που συνδέονται με ναρκωτικά. Αυτό θα επηρεάσει θετικά και τον αριθμό των κρατούμενων και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να θεσπίσουμε και μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα είναι εγγυητής για, ε, για τα δικαιώματα των ε, κρατουμένων και η οποία αρχή θα είναι ήδη λειτουργική από το τέλος Μαΐου η ύπαρξη λοιπόν ενός διαμεσολαβητή για τους κρατουμένους είναι κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας ε, βάσει του πρόσθετου πρωτοκόλου για την πρόληψη των βασανιστήριων των Ηνωμένων Εθνών. 3 Μαΐου 2013 κυρώσαμε αυτή τη σύμβαση και είχαμε ένα χρόνο στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την Εθνική Αρχή Εποπτείας όλων των σοφρονιστικών καταστημάτων της Ιταλίας. Και αυτό είναι μια υποχρέωση που απορρέει από τη ε, δημιουργία αυτής της Επιτροπής στα Ηνωμένα Έθνη. Έχουμε λοιπόν ένα διπλό ρόλο με αυτό το, αυτή τη νέα αρχή διαμεσολάβηση για του κρατούμενους, εσωτερικό ρόλο, μια προσπάθεια να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα και οι διαμάχες στην, ε, στις φυλακές, να υπάρχει νομική υποστήριξη προς τους ε, κρατουμένους και συγχρόνως την ικανοποίηση της δημιουργίας ενός εθνικού προληπτικού μηχανισμού όπως απαιτείται από το προαιρετικό πρωτόκολλο το οποίο εμείς κυρώσαμε των Ηνωμένων Και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς θα εξασφαλίσουμε την υποστήριξη όλων των εταίρων μας στην Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε φυσικά και εμείς από την πλευρά μας έτοιμοι να υποστηρίξουμε όλους τους άλλους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα στις φυλακές τους και όπου υπάρχουν πολλές φορές δύσκολα προβλήματα λόγω υπερπληθυσμού και λόγω της πίεσης που ασκείται από την ε, κοινωνία να αντιμετωπιστούν οι αντιφάσεις στην κοινωνία μας με στέρηση ελευθερία. Ενώ η στέρηση ελευθερία θα πρέπει να είναι μονάχα ένα μέτρο οριστική καταφυγή. Και γι' αυτό ελπίζω ότι κατανοείτε ότι ήταν σημαντική υποστήριξη που δώσατε επισκεπτόμενοι τις φυλακές μας στην Ιταλία και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εργαζόμαστε όλοι ώστε να όχι μόνο να εξασφαλίσουμε την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του, του ΕΔΑΔ αλλά επίσης και ώστε να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε το υπόδειγμα του σοφρονιστικού μας συστήματος στην Ιταλία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πάλμα για την παρουσίαση αυτή και για τις λεπτομέρειες σε σχέση με την πείρα σας και την προηγούμενη ιδιότητά σας. Σας ευχαριστούμε για τις ακόπες προσπάθειες από κοινού μαζί μας για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις και τις δυσκολίες αυτής της κατάστασης. Θα καταλαβαίνετε τι προσπαθούσα να πω όταν μίλησα για το Ποτσορεάλε και την κατάσταση αυτή. Και κυρίως ένα πράγμα τόνισα πάνω απ' όλα. Αυτό αποκόμισα από την επίσκεψή μου στην Ιταλία με τα υπόλοιπα μέλη της Αντιπροσωπείας και την ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα αυτό είναι ότι ναι, υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα, υπάρχουν θεραπείας. Ναι, υπάρχει αυτό το νέο αξίωμα του διαμεσολαβητή για τα δικαιώματα των κρατουμένων, αλλά κάτι λείπει. Μια επιτροπή, μια επιτροπή για τον προπολογισμό που να ανανεώσει τις εγκαταστάσεις των σοφρονιστικών ειδημάτων. Πραγματικά για μένα ήταν ε, πολύ απογοητευτικό ότι το πόντζο Ρεάλε εγκαινιάστηκε το 1910, πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Και αυτό έχει σημασία για, τις, ε, για ένα θεσμικό ίδρυμα όπως μια φυλακή. Οι προδιαγραφέ ε, πριν από 100 χρόνια ήταν τελείω διαφορετικέ από το κράτο δικαίου και τον τρόπο που εμεί αντιλαμβανόμαστε πλέον και που φροντίζουμε για τους κρατουμένους σήμερα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ πραγματικά σας έδωσα εδώ μια Κατάθεση της δικής μου προσωπικής εμπειρίας και εντύπωση ε, ως πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης στην Ισπανία. Ήμουν μέλος της κυβέρνησης. Είχα ορκιστεί, είχα δεσμευτεί να ασχοληθώ με την ανακαίνιση, τέλο πάντων την ανανέωση των σοφρονιστικών ιδρυμάτων στη χώρα μου και να μην συνεχίσουν να λειτουργούν κτίρια ή εγκαταστάσεις που είναι τελείως απριχιωμένες και που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύπτουν τις συνταγματικές απαιτήσεις της νομοθεσίας που άρχισε να ισχύει μετά. Βεβαίως υπήρξαν επικριτικά σχόλια σχετικά, φυσικά υπήρξαν ε, δημαγωγικές και λαϊκιστικές απόψεις εναντίον μου, Ακόμη κάποιοι έφτασαν να πούν ότι οι νέες σοφρονιστικές εγκαταστάσεις έμοιαζαν με πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία. Τα έχω δει και τα έχω διαβάσει σε λαϊκίστικα έντυπα. Όμως το θέμα είναι ακριβώς αυτό, ε, ότι δεν μπορεί να έχουμε 3.000 κατωμένους σε ένα κτίριο το οποίο είναι τελείως ε, υποκατάρρευση. Σκοτεινό, υγρό, φρικτά ζεστό το καλοκαίρι και χωρίς τέρμανση το χειμώνα. Είναι πραγματικά τρομακτικές συνθήκες κράτησης αυτές. θυμίζουν πιο πολύ ε, μυθιστορήματα του 19ου αιώνα και τις περιγραφές τους παρά τις συνταγματικές ε, απαιτήσει και τα πρότυπα που έχουν προβλεφθεί. από το Διεθνές Δίκαιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και κυρίως μέσω των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Κατά κύριο λόγο, με την απαγόρευση στο άρθρο 3 της υποβαθμισμένης μεταχείρισης στην επιβολή ποινών ή τα βασανιστήρια. Διευρύνεται το πεδίο του τι μπορεί να σημαίνει βασανιστήριο σε σοφρονιστικές συνθήκες. Αυτήν την σκέψη όταν την ανέπτυξα στον οποιονδήποτε συνομιλητή μου που συνείδησα δεν είχα κανένα ένδειξη ότι η Ιταλική πολιτική το έθεσε αυτό ουδέποτε ως προτεραιότητα ή τουλάχιστον ως ένα θέμα προσυζήτηση. Ουδέποτε συζητήθηκε η επένδυση, οι επενδύσεις, την ανακαίνιση ή τέλος πάντων την ανανέωση των σοφρονιστικών ιδρυμάτων. Σημαντικές επενδύσεις τελευταίες 20, την τελευταία 20 ετία σε άλλες χώρες, ναι. Πολλά σοφρονιστικά ιδρύματα έχουν γίνει. Ναι, πολλά σοφρονιστικά ιδρύματα και δημιουργήθηκαν και άρχισαν να χρησιμοποιούνται για κράτηση τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια ανάλογα με τις επενδύσεις που έγιναν. Ανάλογα με τις προτεραιότητες που τέθηκαν δηλαδή στον προπολογισμό. Θα θέλατε να το σχολιάσετε αυτό, αλλά ήθελα να δω τι θα πούνε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Νομίζω ο κύριος Μπρόγκς έχει κάτι να πει. Και η κυρία Γκόντς, ως μέλος της αντιπροσωπείας. Θέλετε να πείτε κάτι? Ωραία, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ήταν μια πολύ καλά προετοιμασμένη αντιπροσωπεία. Μάθαμε πολλά από πολλούς εμπειρογνώμονες πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης από τον Υπουργό Δικαιοσύνη μέχρι πολλές οργανώσεις πολιτών που είχαν θέσει ερωτήσεις πολύ σωστές, ε, στοχοθετημένες μέσα σε βραχή χρονικό διάστημα. Όπως ε, είπατε κι εσείς, η κατάσταση ήταν αυτή που περιγράψατε. Η εντύπωσή μου πέραν αυτών ήταν ότι πολλά από τα κοινωνικά προβλήματα στην Ιταλία αντιμετωπίζονται μέσω φυλάκισης. Όπως ξέρουμε, το πρόβλημα στην Ιταλία είναι η μετανάστευση, οι παράνομοι μετανάστες, που τελικά καταλήγουν στις φυλακές και δημιουργούν αυτό τον υπερπληθυσμό των ε, φυλακών. Το άλλο είναι ε, ότι υπάρχει, ε, υπάρχουν τα ναρκωτικά. Και αυτό είναι ένα επιπλέον βάρος για τις φυλακές. Αντί δηλαδή να δημιουργηθεί ένα σύστημα για πρόληψη και θεραπεία, που αυτό καλύπτει μέρος του προβλήματος. Ξέρω ότι συμβαίνει, υπάρχει και πρόληψη και θεραπεία, κυρίως στον ποινικό χώρο, αλλά η εντύπωσή μας είναι ότι ξεπερνούσε τα πλαίσια, ε, αυτά τα πλαίσια και τα, τα ναρκωτικά, δηλαδή οι ναρκωμανείς αντιμετωπίζονται όχι πολύ καλά στις φυλακές. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή, πιστεύουμε, πέραν από τα εναλλακτικά μέτρα που αναφέρατε, θα πρέπει ε, να υπάρχει κουλτούρα σε αυτή τη χώρα. Δεν, ε, οι λύσει δεν μπορούν να δοθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Επίσης πρέπει να δούμε τι γίνεται γύρω μας, ε, να ξεκινήσουν αλλαγές στο σύστημα των κοινωνικών υπηρεσιών και όσον αφορά το, το θέμα των ατόμων που παίρνουν ναρκωτικά, που είναι εθισμένοι στα ναρκωτικά αλλά οι συνθήκες διαβίωσης φυλακές ήταν κάτι το πολύ δυσάρεστο και μόνο η φυσική κατάσταση, αλλά και τα κτίρια υποβαθμισμένα. Η κατάσταση ήταν απαράδεκτη. Αλλά όλο το κλίμα εκεί ήταν δυσάρεστο. Πρωτού φτάσουμε, ή μόλις φτάσαμε, είχε γίνει προσπάθεια, ε, αλλά και ε, υπάρχει καοδιαχείριση όχι μόνο μεταξύ των ε, κρατουμένων αλλά και από το προσωπικό. Το θέμα είναι να περνούν περισσότερο χρόνο εκτός των κελιών τους ε, οι φυλακισμένοι. Είμαι ψυχίατρος και συζήτησα με ορισμένα άτομα που περνάνε 24 ώρες 24 ώρο σε απομονωτήρια και πολλοί από αυτούς είχαν ψυχικά προβλήματα Φυσικά δεν μπορεί να ζει κανεί από αυτά τα συνθήκα και χρειάζεται μία αντιμετώπιση και θεραπεία. Αυτό που είδαμε λοιπόν είναι ένα σύνολο κοινωνικών, ψυχικών προβλημάτων που όλα αυτά συσσωρεύονται μαζί με τον υπερπληθυσμό ε, των κρατουμένων. Ε, δεν μπορούμε με μία λύση να ε, λύσουμε όλα τα προβλήματα. πρέπει η παρέμβαση να είναι πολύμορφη αν θέλετε και πρέπει αυτές οι επισκέψεις να επαναληφθούν διότι γνωρίζουμε ότι στην Ιταλία τα πράγματα είναι δύσκολα αλλά είμαι βέβαιη ότι αν επισκεφθούμε και άλλες χώρες δεν θα βρούμε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ε, από αυτό το κατάλογο των αποτελεσμάτων ε, βλέπουμε ε, από ότι η κατάσταση του δικαστικού σώματος δεν είναι πολύ καλή στην Ιταλία. Πρέπει να βελτιωθεί ώστε να μειωθεί ο χρόνος που περνούν στα κρατητήρια τα άτομα. Ευχαριστώ. Κύριε Μπρόγκς. Σας ευχαριστώ εγώ. Σημείωσα στην παρουσίασή σας από τους 600-828 κρατουμένους, 28.000 περίπου η μισή ήταν ξένοι υπήκοοι από την Τινησία, την Αλβανία και τη Ρουμανία. Με πληροφορούν ότι για τους Ρουμάνους ένας μεγάλος αριθμός είναι από την κοινότητα των Ρώμα. Το ερώτημά μου είναι μήπως είναι αυτό ακόμα ένα σαφές παραδείγμα ε, διάκρισης εναντίον κάποιων εθνοτικών ομάδων. Εάν δεν μπορείτε να εξηγήσετε με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση αυτή, ε, η μόνη άλλη εξήγηση είναι μια εξήγηση η οποία είναι ακόμα χειρότερη, που δεν τολμάει να σπάσει τη σιωπή της, όπως έλεγε ο Όσκαρ Εγώ νομίζω ότι η έκθεση ήταν εντυπωσιακή αλλά και σοκαριστική. Πολλές από τις προτάσεις σας είναι πράγματι λογικές και επικοδομητικές, αλλά ακόμα και το 60% των κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί <clears throat> δεν έχουν καταδικαστεί να ζουν σε απάνθρωπες ανθρώπινες ε, συνθήκες. Επομένως είναι άδικη η μεταχείρισή τους ακόμα και αν έχουν δικαστεί και καταδικαστεί δικαίως. Αναφέρθηκαν βασανιστήρια, κάτι το οποίο με σοκάρει. Δεν μπορούμε να δεχτούμε σε καμία περίπτωση την, τα βασανιστήρια. Αλλά πέραν του σοφρονιστικού συστήματος, οι, τα έχουν χρησιμοποιηθεί από κυβερνήσεις χωρών όπου η, τα βασανιστήρια είναι ποινικό αδίκημα. Ξέρουμε τώρα από αποκαλύψεις ότι και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου του Αντωνίου Μπλερ έχει συνεργαστεί με, τις, ε, με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τις ειδικέ παραδόσεις, για τις έκτασεις παραδόσεις, αλλά ξέραν ότι αυτό θα οδηγήσει σε βασανιστήρια. Όλοι λοιπόν οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων που ε, συγκαλύπτουν τα βασανιστήρια αυτά θα πρέπει να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης αλλιώς τα θέματα αυτά δεν θα μπορέσουν ποτέ να αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ κύριε Μπρόγκος για επικοδομητικά σας <clears throat> συμπεράσματα. Σας πω όμως το εξής. Τα θέματα των βασανιστήριων έχουν τονιστεί πολλές φορές και σε ανταλλαγές απόψεων με πολλούς συνομιλητές μας και αυτό περιλαμβάνει και τις ε, δύο νομοθετικές συνελεύσεις. Μάθαμε λοιπόν ότι αντίθετα από τις περισσότερες νομικές ρήτρες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ιταλική Δημοκρατία έχει ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος μέχρι τώρα που δεν θεωρεί ως ε, συγκεκριμένο αδίκημα το αδίκημα της, ε, των βασανιστήριων. Κάτι λοιπόν το οποίο θα έδινε λαβή σε, σε μηνύσεις εναντίον των ε, σε καταγγελίες εναντίον των σοφρανιστικών υπαλλήλων που θα, θα ασκούσαν βασανιστήρια στους κρατουμένους. Για να μπορέσουν λοιπόν να διωχθούν αυτά τα αδικήματα μπορούν μονάχα να καταγγελθούν ως κατάχρηση εξουσίας αλλά όχι συγκεκριμένα ως βασανιστήρια. Μας πληροφορήσανε ότι γίνονται βέβαια μεταρρυθμίσεις, ότι υπήρξε μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για να καλυφθεί αυτό το νομικό κενό σε άλλες χώρες τα βασανιστήρια μπορούν να διωχθούν και μπορεί να προκύψει δικαστική διαδικασία ακριβώς λόγω μιας καταγγελίας βασανιστήριων. Εναντίον ενός σοφρανιστικού υπαλλήλου, ενός δεσμοφύλακα, ενός αξιωματούχου των φυλακών που εφαρμόζει τέτοιου είδου βασανιστήρια στους κρατουμένους. Αλλά αυτό το είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν οι υλικέ συνθήκες στις φυλακές ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμόζονται τα πρότυπα που αναφέρει η απόφαση του, ΕΔΑΔ. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστούν οι, ειδικές, οι υλικές αυτές συνθήκες. Το Πότζιο Ρεάλε είναι πραγματικά ένα αρνητικό παράδειγμα γιατί όλη η δομή του κέντρο αυτού είναι να μένουν οι κρατούμενοι ώστε τέτοια που να κάνει τους κρατουμένους να είναι συνέχεια μέσα στα κελιά τους και είναι αφόρτη η κατάσταση λόγω του υπερπληθυσμού της φυλακής. Όταν είναι συνέχεια λοιπόν κλειδωμένοι οι κρατήροι, οι κρατούμενοι, αυτό δεν έχει μονάχα αφόρτες συνέπειες για τους ίδιους, αλλά όταν το βλέπει κανείς και με τα μάτια του, αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει να καταλάβουμε πόσο απάνθρωπα είναι όλα αυτά. Εγώ εθλίβην βαθύτατα. Βλέποντας ότι μόναχα και αν είχαμε μεταφέρει αυτούς τους κρατουμένους σε κάποιο άλλο κέντρο, θα σταματούσαν οι συνθήκες κράτησης να είναι τόσο επιθετικά απάνθρωπες όπως αυτές που είδαμε στο Πόζιο Ρεάλε. Και το λέω με κάθε σεβασμό βέβαια, για, τον, ε, για τις προσπάθειες της Ιταλικής κυβέρνησης και την προσωπική δέσμευση των επικεφαλής της φυλακής, οι οποίοι κάνουν το καθήκον τους εφαρμόζουν το ποινικό δίκαιο της ε, Ιταλίας, αλλά είναι μια πραγματικά αντικειμενική κατάσταση ότι το κτίριο αυτό μαζί με τον υπερπληθυσμό δεν μπορεί να είναι συμβατό με τα ανθρώπινα πρότυπα για την κράτηση φυλακισμένων και με την κατανόηση του πώς θα πρέπει κανείς να εκτίσει μία ποινή στέρησης της ελευθερίας. Επανερχόμαστε λοιπόν στον κύριο Πάλμε, αν θέλει να κάνει κάποια σχόλια, θέλετε να πείτε κάτι. Δύο ή τρία σύντομα σχόλια. Πρώτα απ' όλα, για το έγκλημα των ε, βασανιστήριων στο δικό μας ποινικό κώδικο, κώδικα. Και αυτό είναι ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί ως το δυνατόν συντομότερα. Διότι μιλήσατε και για τη σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστήριων πριν από μία εικοσαετία. Και πρέπει να πω ότι το θέμα είναι πώς κρίνουμε ε, την μεταχείριση των κρατουμένων αλλά χωρίς την κατηγορία ή το αδίκημα των βασανιστήριων με μια απλή ε, κατάχρηση, επίθεση με με κάποιο άλλο είδους ε, σωματικές βλάβες, αυτό είναι πολύ εύκολο να ε, απαλληφθεί τελείως, να παραγραφεί. Καθαρίζεται εφόσον υπάρξει όμως καλή εκδίκαση και ε, εφόσον η Βουλή μας εγκρίνει το νόμο που εξετάζει η Γερουσία, ελπίζω ότι το κενό αυτό θα καλυφθεί στο προσεχές μέλλον. Ένα άλλο ζήτημα που αναφέρθηκε είναι το αρχιτεκτονικό σχέδιο ή τέλο πάντων πολεοδεμικά πώς έχουμε σχεδιάσει τις φυλακές μας. Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός των χώρων είναι ενδεικτικός όντως του βίου που μπορεί κανείς να διάγει σε ένα τέτοιο χώρο. Σε ένα χώρο λοιπόν που έχει σχεδιαστεί σε μια τιμωρητική αντίληψη όπως ε, κυκλοφορούσε πριν από 100 χρόνια, ναι, είναι πολύ δύσκολο σήμερα να έχει την οποιαδήποτε εγκυρότητα. Έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη περί κράτησης σήμερα. Οπότε ναι, υπάρχει ανάγκη να, επενδύσουμε στην ε, ανακαίνιση, την εκβάθρον ανακαίνιση των ιδρυμάτων μας. Αυτό δεν θα είναι απλό, ιδίως σε μια περίοδο κρίσης, όπου η στήριξη και συμφωνία της υπόλοιπης κοινωνίας είναι πολύ χαμηλή, αλλά είναι κάτι που πρέπει να τεθεί επιτάπητος και να προωθηθεί στις πολιτικές μας συζητήσεις. Αυτό συνδέεται άμεσα και με το άλλο ζήτημα, με το θέμα των κοινωνικών υπηρεσιών θα πρέπει να ξανασχεδιάσουμε αυτό το σύστημα έχοντας υπόψη ότι η κράτηση, η φυλάκιση είναι ένα μέρος του συστήματος. Δεν είναι κάτι που πρέπει να, απομπε... να απεμβολήσουμε από το υπόλοιπο σύστημα. Δεν είναι ένα τμήμα τελείως αυτόνομο. Γι' αυτό η στήριξη των εταίρων μας στην Ευρώπη είναι απαραίτητη και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι κάποιοι από τους κρατούμενου που διαμένουν στις φυλακές μας, που κρατούνται στις φυλακές μας, μπορεί να είναι πολίτες άλλων κρατών μελών. Ξέρετε πώς ε, ε, επίπεδα προστασίας υπάρχουν για τους αλλοδαπούς ε, στα φροντικά ιδρύματα οικίας χώρας. Υπάρχει μια κατηγορία για τους πολίτες ευρωπαϊκών κρατών. Μια άλλη κατηγορία για τις χώρες των, του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπόκεινται στα όσα ορίζει η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και μετά υπάρχουν και πολίτες άλλων, τρίτων χωρών, που δεν είναι μέλη ούτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οπότε αυτές τις τρεις κατηγορίες πρέπει να τις έχουμε διαρκώ υπόψη. Για όσου είναι πολίτε τη Ένωση. Εκεί πρέπει να έχουμε τη βοήθεια των εταίρων μας για να μπορούμε να τους μετακινήσουμε στις ε, οικίες εθνικές τους φυλακές. Για όσους είναι πολίτες χώρας Συμβουλίου της Ευρώπης θα πρέπει να μπορεί να γίνει το ίδιο. Δεδομένου ότι καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για όσους μπορεί να είναι από χώρες όπως το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τινησία. Η κατάσταση διαφέρει, διότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί και να ε, είμαστε πιστοί στην αρχή της μη επαναπρόθεσης. Πρέπει να υπάρξουν διμερείς συμφωνίες ώστε να προβλέπεται και δυνατότητα οι άνθρωποι αυτοί να μετακινηθούν αλλά υπό συνθήκες ασφάλειας είναι περίπου οι αδρές γραμμές της δικής μας δράσης. Δεν έχω καμία επιλογή παρά να συμφωνήσω απολύτως με τη δική σας αποτίμηση για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που σημειώσατε κατά την επίσκεψή σας. Πρόεδρος, εκτός... Χωρίς μικρόφωνο, πρόεδρος. Έχοντας ακούσει λοιπόν και τις απόψεις των μελών, Θέλει κάποιος να σχολιάσει τα θέματα αυτά από την Κομισιόν για την έκθεση, αν θέλετε να είστε σύντομος. Η Ελληνική Προεδρία, επίσης, κανένα σχόλιο από εμάς. Ευχαριστώ. Ούτε η Κομισιόν. Ούτε και εγώ έχω σχόλια, κύριε Πρόεδρε. Ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. γιατί υπάρχει πρόβλημα αποτελεσματικότητας και υπάρχει των νομικών θεραπείων και λόγω αυτών ένα αχανές τμήμα του πληθυσμού των φυλακών δεν είναι εκεί επειδή είναι καταδικασμένοι αλλά είναι πολλές φορές προφυλακισμένοι και είναι εκεί λόγω των καθυστερήσεων του δικαστικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διάφορα κράτη-μέλη. Αλλά φυσικά υπάρχουν και ιδιαιτερότητε στην Ιταλία που είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε η διεισόμαση και πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο ψηφίσματος, το σχέδιο έκθεσης θα καταδείξει την, ε, το πρόβλημα αυτό και την ανάγκη να δοθεί συνέχεια από το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Περνάμε λοιπόν στο τελευταίο σημείο σήμερα Πρόκειται για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα θέματα προσωπικών δεδομένων. Υπήρξε λοιπόν αυτή η απόφαση που δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο νοιάζεται για τα προσωπικά δικαιώματα και τα προσωπικά στοιχεία των Ευρωπαίων πολιτών για το κράτος δικαίου, για την ασφάλεια δικαίου, για τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στη συνθήκη της Λισαβόνας με την συμπερίληψη της Χάρτας ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αλλά όλα αυτά μας θυμίσουν και πάλι ότι υπάρχει μια ανάγκη, μια κατεπίγουσα ανάγκη για να ενημερώσουμε, να επικαιροποιήσουμε το σύστημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη. Υπογραμμίζει την αναγκαιότητα και το κατεπήγον του να αποφασίσει το Συμβούλιο σε σχέση με το πακέτο για την φύλαξη προσωπικών δεδομένων και την οδηγία και τον κανονισμό γιατί μια κοινή θέση του Συμβουλίου θα σηματοδοτούσε την πολιτική θέληση να συζητήσει και να διαπραγματευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια τέτοια επικαιροποίηση η οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσει να ενισχύσει τον ιδιωτικό χαρακτήρα των δεδομένων και την ασφάλεια δικαίου για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλουμε λοιπόν να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό το θέμα, για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 8ης Απριλίου, που αποφάσισε ότι η οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα του 2006 παρεμβαίνει στα προσωπικά δικαιώματα και την προσωπική ζωή και έχουμε εδώ την ε, ε, νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα παρουσιάσει αυτή την απόφαση και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Κύριε Καγιόλα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην απόφαση του, της 8ης Απριλίου 2014 που έπεται των αποτελεσμάτων του κ. Βίζα υπό την ίδια έννοια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεώρησε ως άκυρη την οδηγία για τη διατήρηση των δεδομένων τα οποία είναι αντικείμενο επεξεργασία στα πλαίσια της παροχής ηλεκτρονικών στοιχείων στο κοινό. Αυτή η απόφαση ε, είναι η συνέχεια δύο ε, προδικαστικών αποφάσεων της High Court της Ιρλανδίας και του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας. Οι δύο υποθέσεις αντιμετωπίστηκαν από κοινού. Το, βασι... Ο βασικός στόχος ε, της οδηγίας αυτής είναι να αρμονίσει τις διατάξεις των κρατών μελών όσον αφορά τη διατήρηση ορισμένων δεδομένων που παράγονται ή γίνονται ε, αντικείμενα επεξεργασία από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή από δημόσια δίκτυα επικοινωνιών. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα για την έρευνα, την πρόληψη, την ανείχνευση και ε, την αντιμετώπιση σημαντικών ποινών, κυρίω του οργανωμένου εγκλήματο και τη τρομοκρατίας. Οι πιο αμφιλεγόμενε διατάξει είναι εκείνες που έχουν σχέση με την υποχρέωση διατήρηση των δεδομένων, την πρόσβαση στα δεδομένα, ε, τι κατηγορίε των ε, δεδομένων που θα διατηρηθούν, τη διάρκεια διατήρηση φύλαξη και την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων. Η οδηγία για φύλαξη των δεδομένων υπήρξε αντικείμενο ε, προσφυγή, την οποία έχουμε λησμονήσει, υπόθεση SIT 301 06 Ιρλανδίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου, αλλά τότε είχε απορριφθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτή η προσφυγή με την απόφαση της 10 Φεβρουαρίου 2009. Αυτή η υπόθεση αφορούσε μόνο τη συζήτηση επιστημονικη βάσης. Με αυτές τις προδικαστικές υποθέσεις, τι οποίες συζητούμε σήμερα, η Ιρλανδική και Αυστριακή Δικαστική Αρχή έθεσαν πολλά θέματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που αφορούσαν και την εγκυρότητα και την ερμηνεία της οδηγίας. Το δικαστήριο επικεντρώθηκε στα θέματα που αφορούσαν την εγκυρότητα της οδηγίας σε σχέση με τα άρθρα κυρίως 7 και 8 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς υπόμνησή σας, το άρθρο 7 της Χάρτας αφορά την, ε, το σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το άρθρο 8 αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Καταρχήν, το δικαστήριο επενθύμησε ότι η υποχρέωση που επιβάλλεται από τα άρθρα 3 και 6 της οδηγίας στους παρόχους υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών ηλεκτρονικής μορφής να διαφυλάξουν ε, για ορισμένο χρονικό διάστημα τα δεδομένα που έχουν σχέση με την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου αποτελεί αφεαυτή σε μια παρεμβολή ε, στα δικαιώματα που προβλέπει το άρθρο 7 της Χάρτας. Επίσης, η πρόσβαση των αρμοδίων εθνικών αρχών στα δεδομένα είναι μια επιπλέον παρεμβολή ε, στα θεμελιώδη δικαιώματα. Επίσης, η οδηγία αποτελεί η ίδια παρεμβολή στο θεμελιώδη δικαίωμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων που εγγυάται το άρθρο 8 της χάρτας. Συνεπώς ε, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι αυτή η παρεμβολή που έχει σχέση με το θεμελιώδη δικαίωμα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της χάρτας είναι μεγάλη έκταση και θα πρέπει να εκλειφθεί ω ιδιαίτερα σοβαρή. Το δικαστήριο επίσης υπογράμμισε ότι ότι οι προποθέσει διαφύλαξης των δεδομένων και η μεταγενέστερη χρησιμοποίηση αυτών των δεδομένων γίνονται χωρί ο χρήστη να έχει ενημερωθεί. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ε, για τα άτομα τα οποία φύγονται ε, το συνέστημα ότι η ιδιωτική του ζωή παρακολουθείται συνέχεια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η διαφύλαξη αυτών των δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί ως ικανή να πραγματοποιήσει το στόχο που επιδιώκεται από την οδηγία. Αλλά αναφορικά με τον, τον απαραίτητο χαρακτήρα διαφύλαξη των δεδομένων, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ο στόχος της καταπολέμησης του σοβαρού εγκλήματος, κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, δεν μπορεί να δικαιολογήσει ένα μέτρο διαφύλασης όπως εκείνη που προβλέπεται από την οδηγία να θεωρείται ως αναγκαία. Το δικαστήριο συνεπώς θεώρησε ότι θα έπρεπε να πιστοποιήσουμε την αναλογικότητα, αναλογικότητα επαναλαμβάνω, της διαπιστωμένης παρεμβολής. Η αρχή της αναλογικότητας απαιτεί όπως οι πράξεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ικανές να πραγματοποιήσουν τους νόμιμους επιδεκόμενους στόχους από την σχετική νομοθεσία και να μην ξεπερνάει τα όρια του καταλήλου και απαραίτητου για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι σε αυτή την περίπτωση και αυτό ήταν αντικείμενο μεγάλη συζήτηση στο δικαστήριο λόγω του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λαμβάνοντα υπόψη τη έκταση και τη σοβαρότητας τη παρεμβολή ε, τη οδηγία επ' αυτού, η εκτίμηση του νομοθέτη περιορίζεται και υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο. Πράγματι, Αναφορικά με το δικαίωμα για προστασία προσωπική ζωή, η προστασία αυτού του θεμελιώδου δικαιώματο απαιτεί σύμφωνα με την ομολογία του Κωστηρίου παρεκκλήσει από την προστασία των προσωπικών δεδομένων να υπάρχουν στα πλαίσια του απαραίτητου. Ο, η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπώ, θα πρέπει να έχει σαφεί κανόνε, επιβάλλοντα μεταξύ άλλων ελάχιστε απαιτήσει προκειμένου τα άτομα των οποίων τα δεδομένα έχουν διαφυλαχθεί να διαθέτουν επαρκείς εγγύησης ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά τα προσωπικά τους δεδομένα έναντι ε, του κίνδυνου κατάχρησης και κάθε παράνομη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η οδηγία διαφύλαξη των δεδομένων επιβάλλει την διατήρηση όλων των σχετικών των δεδομένων που έχουν σχέση με τη σταθερή τηλεφωνία, την κινητή τηλεφωνία, την πρόσβαση στο διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω διαδικτύου καθώ και τηλεφωνία μέσω διαδικτύου. Αυτή η οδηγία καλύπτει γενικά κάθε άτομα και όλα τα μέσα επικοινωνίας ηλεκτρονικής καθώς και το σύνολο των δεδομένων που έχουν σχέση με αυτή τη διακίνηση χωρίς καμία διαφοροποίηση, περιορισμό ή εξαίρεση ανάλογα με το στόχο της καταπολέμησης των σοβαρών εγκλημάτων. Επίσης, η οδηγία δεν απαιτεί καμία σχέση ανάμεσα στα δεδομένα των οποίων προβλέπεται η διαφύλαξη και μια άμεση απειλή για την δημόσια ασφάλεια. Επίσης δεν περιορίζεται σε διαφύλαξη που αφορά είτε ε, δεδομένα που έχουν σχέση με μια μεταβατική περίοδο είτε μια καθορισμένη γεωγραφική ζώνη. Επίσης η οδηγία δεν προβλέπει και η πρόσβαση και η μεταγενέστερη χρήση των δεδομένων αυτών να περιορίζεται μόνο για ε, την πρόληψη, την ανείχνευση σοβαρών εγκλημάτων, που κατονομάζονται ρητά. Πράγματι, το άρθρο 4 της οδηγίας περιορίζεται να προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος ε, αποφασίζει για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για να υπάρχει πρόσβαση στα διατηρούμενα δεδομένα ε, σεβόμενη τις απαιτήσει, τις ανάγκες και αναλογικότητας χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Υπογραμμίζει επίσης το δικαστήριο ότι η πρόσβαση στα διατηρούμενα δεδομένα από τις εθνικές αρχές, αρμόδιες εθνικές αρχές, δεν υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο που διενεργείται είτε από τις δικαιοδοτικές αρχές, είτε από μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Επίσης, το δικαστήριο υπογραμμίζει ότι η οδηγία επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων για ένα εξάμεινο χωρίς διάκριση μεταξύ κατηγοριών δεδομένων. Επίσης, η διάρκεια της διατήρησης είναι μεταξύ 6 μηνών το ελάχιστο και 24 μηνών το μέγιστο, χωρίς αντικειμενικά κριτήρια να έχουν διευκρινιστεί προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η διατήρηση αυτή περιορίζεται στο απαραίτητο. Για μία ακόμη φορά, ε, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογικότητα. Καταλήγει λοιπόν το δικαστήριο ότι η οδηγία δεν προβλέπει σαφείς κανόνες που διέπουν την έκταση και την παρέμβαση στα εθνικά δικαιώματα που ορίζουν τα άρθρα 7 και 8 της χάρτας. Το δικαστήριο θεωρεί ότι η μεγάλη παρεμβολή στα ε, θεμελιώδη δικαιώματα δεν περιβάλλεται από τις διατάξεις που επιτρέπουν να διασφαλίζεται ότι αυτή η παρέμβαση πράγματι περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο. Τέλος, το δικαστήριο παρατηρεί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι σε σχέση με τους κινδύνους παράνομης πρόσβασης, η εχεμήθεια των δεδομένων δεν διασφαλίζεται και δεν υπάρχει υποχρέωση που να εξασφαλίζει ότι αυτά τα δεδομένα διατηρούνται μόνο στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, το δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η οδηγία παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και συνεπώς θεωρείται ακυρή στο σύνολό της. Αυτή η δήλωση ακυρότητας δεν φύγει αυτή την πράξη, αλλά αυτή η πράξη που θεωρείται άκυρη έχει αναδρομική ισχύ, όπως συμβαίνει με την οδηγία που συζητούμε πέραν. Οι δικαστές θα πρέπει να θεωρήσουν ότι αυτή η πράξη είναι άκυρη για τις ανάγκες ε, μιας απόφασης την οποία θα εκδώσει και η εθνική δικαιοδοσία δεν μπορεί πλέον να εφαρμόσει αυτή την πράξη που θεωρείται άκυρη. Οι εθνικές πράξεις και η μεταφορά της οδηγίας δεν ε, ακυρώνονται, αλλά εναπόκειται σε εθνικές δικαιοδοσίες αρχές να αποφανθούν για την εγκυρότητά τους. Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να παρουσιάσω μια σύνθεση των ε, αποφάσεων του δικαστηρίου. Σίγουρα αυτή η απόφαση γύρει πολλά ερωτήματα. Η νομική υπηρεσία αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των θεμάτων και αναφέρει απλώς και σε εσά και στην Επιτροπή ότι είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα αφού γίνει μια εις ανάλυση η οποία είναι απαραίτητη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Καγιόλα. Τονίζετε ότι στις αποφάσεις του το δικαστήριο ακολούθησε το, την άποψη του πρώην συνταγματικού δικαστηρίου της Ισπανίας, του κυρίου Μαγιόλ, διότι σε θέματα συνταγματολογικά και χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Είχαμε και έγκριση της οδηγίας αυτή μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001, το 2004 στην Ισπανία, 2006 στο Λονδίνο και το αποτέλεσμα είναι ότι η οδηγία δεν συνάδει με το επίπεδο προστασίας του ιδιωτικού βίου και τη θέση σε ισχύ της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Μας θυμίζει την ανάγκη να συμπληρωθεί το νομοθετικό πακέτο σε προστασία των δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων, πιο συγκεκριμένα της οδηγίας. Διότι η οδηγία καλείται να ε, εξασφαλίσει την ασφάλεια των δημόσιων φορέων, των ε, κρατικών ε, λειτουργών, των διοκτικών δυνάμεων, των ε, κρατικών ερευνών και ανακρίσεων μετά από ύποπτες κινήσεις, υποψιών συμμετοχής ατομοκρατική οργάνωση. οι υποψίες για απειλές κατά της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών, για αυτό που να συμπληρωθεί το νομοθετικό πακέτο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή ένας νέος κανονισμός και μια νέα οδηγία είναι απαραίτητα. Τώρα ακόμα έχουμε λίγα λεπτά για συζήτηση. Και μετά, finalement, il y να ακούσουμε τους συναδέλφους και μετά ίσως να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πρόεδρο ΡΕΚ. Ο κύριος Φως, έχετε πρώτος το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι γνωρίζω, είναι δύο σημεία τα οποία γίνονται σαφή με αυτή την απόφαση ότι γενικά μπορεί να υπάρξει φύλαξη δεδομένων προσωπικών, αλλά εάν υπάρχει εγγύηση της αναλογικότητας από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, δεν πρέπει να καταλήξει κανείς το συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία φύλαξη προσωπικών δεδομένων, όχι δεν πρόκειται περί αυτού. Απλώς πρέπει να αλλάξουμε την τωρινή οδηγία, γιατί η δική μας ευθύνη είναι να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των θεμητών συμφερόντων των πολιτών για να προστατευτούν τα προσωπικά του δεδομένα από τη μία πλευρά, αλλά συγχρόνως έχουν θεμητό συμφέρον να υπάρχει και η διερεύνηση σοβαρών αδικημάτων. Και εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια διαδικασία δίωξη η οποία βασίζεται όλο και περισσότερο σε ανάλυση δεδομένων. Επομένω, θα πρέπει να δίνεται τη δυνατότητα στι διοικητικέ αρχέ να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Βέβαια, ο νομοθέτης θα πρέπει να εξασφαλίσει και όρια, να είναι δυνατόν δηλαδή να γίνεται αυτή η δίωξη της εγκληματικότητος που βασίζεται σε, η δίωξη αυτή που βασίζεται σε δεδομένα και να μην δίνεται η δυνατότητα στους εγκληματίες να διαφεύγουν. Από την άλλη πλευρά, πέραν της ε, ανάγκης ενός κράτους να διώχνει την ε, ε, εγκληματικότητα πρέπει να εξασφαλίσει και την προστασία των θυμάτων τέτοιων εγκλημάτων, δηλαδή όλα αυτά είναι μια κρατική αρμοδιότητα για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και στους ε, οικίους των θυμάτων εάν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα, γιατί δεν μπορούμε να διαλευκάνουμε πλήρως μια εγκληματική πράξη. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν θεσπίζουμε τα όρια στη χρήση των προσωπικών δεδομένων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Είναι όλα αυτά λοιπόν στοιχεία τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητα για τον κολασμό των σοβαρών εγκλημάτων και δεν θα πρέπει να μειώσουμε τις προσπάθειές μας να υποστηρίξουμε τις διοκτικές αρχές ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα θέματα γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο αυτοδικίας όταν λέμε ότι για λόγους προσωπικών, προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν θα μπορούμε να διερευνήσουμε πλήρως ορισμένα αδικήματα. Τι θα κάνει τότε ο απλός πολίτης όταν έρθει αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα σωστό πλαίσιο το οποίο θα μπορέσει να εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη σε σχέση με αυτά τα ε, δεδομένα. Ευχαριστούμε κύριο Μωράης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Επειδή λέμε το πώς αισθανόμαστε για την απόφαση, αλλά όχι μόνο, να ρωτήσω την νομική υπηρεσία. Τι γίνεται με την αναδρομική ισχύ της απόφασης. Μπορείτε να μου το διευκρινίσετε. Τι σημαίνει σε εθνικό επίπεδο για τις εθνικές νομοθεσίες αυτό. Για τις εθνικές νομοθεσίες. Τι γίνεται με τη φύλαξη δεδομένων αυτή τη στιγμή από τα κράτη-μέλη. Τα δεδομένα που ήδη δηλαδή ε, φυλάσσονται και πώς θα μπορούν να ανακαλούνται οι νόμοι για την ε, φύλαξη. Δεν ήταν πολύ σαφές και αυτό το θέμα γίνεται όλο ένα και πιο σοβαρό. Αν διαβάζει αν διαβάζει κανεί την υπόθεση, δεν είναι τελείως σαφέ πώ θα διευθετηθεί αυτό και θα ήθελα σε από την νομική υπηρεσία. Ω προς την ε, σημασία, το νόημα τη απόφαση αυτή. μπορούμε να την αναγνώσουμε και προσπαθούμε να την κατανοήσουμε, αλλά ω τώρα η κατανόησή μας λέει το εξή, Είναι μια απόφαση αρκετά συστηματική γιατί στέκεται σε κάθε διαφορετικό στοιχείο ξεχωριστά ως προς την ε, αναλογικότητα, την ε, ανεπάρκεια των ε, στοιχείων, την πρόσβαση. Αυτά είναι στη σημεία που είχαμε συζητήσει και βάσει της αρχικής πρότασης πριν από δυόμιση χρόνια και η οδηγία για την φύλαξη δεδομένων είχε αρχίσει να συζητιέται όταν ως ομάδα στηρίζαμε την πρόταση αυτή. Όμως θεωρούσαμε ότι χρειάζεται μια προεδραστική έγκριση λόγου χάρη. Τελικά κάθε σημείο της απόφασης αυτής είναι κρίσιμη σημασία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η απόφαση είναι σημαντική και το σκηνικό από εδώ το που συζητιέται την πρόταση αυτή έχει αλλάξει τελείως. Αυτό που πλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι κάτι σαν ε, ένα, μια κλίση να ξυπνήσουμε και να δράσουμε. Σίγουρα είναι σαφές πια ότι χρειάζεται κάποια φύλαξη δεδομένων και σίγουρα χρειάζεται και προστασία τους. Υπάρχουν απειλέ κατά τη ασφάλεια, υπάρχουν τρομοκρατικέ απειλέ και εκεί τα δεδομένα χρειάζονται. Προ την αναλογικότητα όμω ή τον κίνδυνο τη παράνομη πρόσβαση, σίγουρα δεν είναι ο καταλληλότερο τρόπο αυτό που έχει ω τώρα επιλεγεί. Αν δείτε κάποια παραδείγματα από την απόφαση, λόγου χάρη, εκεί που γίνεται λόγο για την τήρηση των δεδομένων από ένα εξάμεινο με μέγιστο όριο δύο χρόνια, αλλά χωρί κατηγοριοποίηση. Η απόφαση αυτή κανονικά είναι πολύ συστηματική. Και το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να συλλέγονται και να κρατώνται, να τηρούνται τα δεδομένα χίδιν όπως γινόταν ως τώρα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχει διευθετήσει η απόφαση. Και το επόμενο που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι ως Κοινοβούλιο ψηφίσαμε την οδηγία και τον κανονισμό ως πακέτο, αλλά θα πρέπει πριν ψηφιστούν αυτά να αποκριθεί και το, το Συμβούλιο. Διότι εμείς τη δική μας τη θέση την εκφράσαμε και έπειτα ίσως να υπάρχει περιθώριο για κάποια επιπλέον νομοθεσία, για να δούμε πώς ακριβώς θα γίνεται η τηρήση των δεδομένων για την αντιμετώπιση των ε, τρομοκρατικών απειλών για θέματα ασφαλείας δεδομένα για αυτά ίσω να πρέπει να μπουν σε μια ειδική κατηγορία. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να καλέσουμε το Συμβούλιο να απαντήσει στην οδηγία που υπάρχει. Και αυτό δεν το κάνουν καθόλου. Και δεν το κάνουν σε καμία περίπτωση γρήγορα. Το θέμα λοιπόν είναι να αναγνωρίσουμε ότι η απόφαση αυτή είναι καταστρεπτική επί οποιασδήποτε διάστασης και αν την πιάσει κανείς και Θέλω πραγματικά να τα σημειώσετε τα σχόλιά μου για το θέμα, γιατί η απόφαση είναι σοβαρή. Είναι σοβαρή και με την ε, τεχνολογία που μεταλλάσσεται διαρκώ, μεταβάλλεται διαρκώ, με την νομοθεσία που χρειαζόμαστε για τι απειλέ κατά τη ασφαλεία μα, ε, σίγουρα κάτι χρειάζεται, αλλά εδώ τα πράγματα πρέπει να κρυθούν. Ναι, αλλά πλησιάζουμε προς το τέλος της πρωινής μας ε, συνεδρίασης. Οπότε θα παρακαλέσω τους συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο να παραμείνουν σύντομοι για να προλάβουμε να ακούσουμε και την Επιτροπή και το Συμβουλίο. Κυρία Σαρχεντίνη, ευχαριστώ Πρόεδρε, κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε την εντύπωση ότι μπορούμε να τα προλάβουμε όλα στο τέλος μιας θητείας όπως θα υποψιάζεται ο καθένας. Αυτή την αντίποση έχω, αλλά εδώ γύρεται μια σειρά από ερωτήματα. Εάν κατάλαβα καλά το δικαστήριο δηλώνει ότι η οδηγία αυτή δεν θα έπρεπε να είχε υπάρξει χωρίς αναδρομική ισχύ. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί. Τι συμ... Θέλω να ρωτήσω την νομική υπηρεσία τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την κάθε εθνική νομοθεσία. Στη δική μου την ε, χώρα τα δεδομένα ε, ήδη συλλέγονται και κρατώνται. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα μας χρειαστεί κάποιο διάστημα να μελετήσουμε την απόφαση βέβαια, αλλά πρέπει μετά να διεξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Σημαίνει για το δικαστήριο, αυτό που λέει το δικαστήριο, ότι δεν έχουμε δικαίωμα να τηρούμε οποιαδήποτε δεδομένα. Και όπως είπε και ε, μια σουηδική εταιρεία στο διαδίκτυο, δεν θα κρατούμε καθόλου δεδομένα γιατί αυτό λέει το δικαστήριο από εδώ και μπρος. Προβλέπω λοιπόν ότι στο προσεχές μέλλον θα υπάρξουν αρκετά προβλήματα με την απόφαση. Τι σημαίνει ως προς την τήρηση δεδομένων των τελευταίων ετών, τι θα γίνει με αυτά που ήδη φυλάσσονται. Και τι γίνεται με ένα μονομοθέτημα που ξαφνικά ακούμε ότι δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει. Και θα υπάρξει και αναδρομική ισχύ στην απόφαση. Τι σημαίνει για τη συμφωνία για τα Μητρώα Επιβατών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς θα επηρεαστούν οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τήρηση αρχείων των ονομάτων των επιβατών λόγου χάρη. Θα επιτρέπονται αυτά ή όχι. Διότι εγώ θεωρούσα ότι η φύλαξη δεδομένων δεν επιτρέπεται αυτήν την έννοια. Οπότε, Επιτροπή, τι θα κάνετε με τα κράτη-μέλη, διότι Ίσως να προκύψουν διαδικασίες επί παραβάση για τα κράτη-μέλη. Διαδικασίες βάσει του νόμου που εντωμεταξύ όμως το δικαστήριο τον έχει ε, κηρύξει άκυρο. Λέει ότι δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει. Πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά. Δεν το βρίσκω καθόλου συνετό να περιμένουμε την επάνωδο του Κοινοβουλίου, δηλαδή την επόμενη θητεία για να απαντηθούν τα θέματα αυτά, διότι όσοι αυτή τη στιγμή φυλάσσονται από εταιρείε τηλεπικοινωνιών, αεροπορικέ εταιρείε, από παρόχου, από οποιονδήποτε, μπορεί πλέον να είναι παράνομα. Θα γίνει ένα, μια έκρηξη εκδίκαση υποθέσεων στο κάθε κράτο μέλο. Ο καθένα θα κοιτάζει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να καταγγείλει. Οι πολίτε μπορούν να διεκδικήσουν το δικαίωμα να μην τηρούνται πια τα δεδομένα τους, οπότε θα ήθελα να μου πει και ο κύριος Φως. Πότε, κατά την άποψή του, είναι ένα αδίκημα αρκετά σοβαρό ώστε να δικαιολογείται η τήρηση δεδομένων. Δεν υπάρχει μια σαφής ορισμός εδώ, όπως ξέρετε, και καλό θα ήταν τέτοιοι ορισμοί να προκύψουν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μόνο ένα σύντομο ερώτημα θέλω να σας θέσω σε σχέση με αυτή την απόφαση. Τα τελευταία δέκα χρόνια που μας απασχολεί το θέμα αυτό των προσωπικών δεδομένων αναρωτιέμαι ποια είναι η διαδικασία που θα μπορούσε να ακολουθηθεί σε μια τέτοια περίπτωση αν υπάρξει μια προσφυγή επί παραβάση χάρη πόσο μπορεί να έρθει ενώπιον των δικαστηρίων το θέμα αυτό της ε, ακύρωσης των εθνικών <clears throat> προτύπων. Γιατί αυτό έχει προκύψει σε σχέση με ένα κράτος μέλος. Αν εξακολουθεί λοιπόν να ισχύει κάποια νομοθεσία ε, και δεν έχει τηρηθεί, τι γίνεται. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θα υπάρξει κάποιο, κάποια προθεσμία για να τροποποιηθεί η εθνική νομοθεσία η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τι θα γίνει στα, στα δικαστήρια, τι θα γίνει με τα δεδομένα τα οποία έχουν ήδη συλλεγεί βάσει εθνικών αποφάσεων, πώς μπορεί κανείς να ε, προσβάλλει αυτές τις αποφάσεις, ποιος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει αγωγή εναντίον αυτών των αποφάσεων, ή η κομισιον ή κάποιος άλλος. Κύριος Μπρόγκς και μετά η Κομισιόν και η Ελληνική Προεδρία. Παρακαλώ. Αν θέλετε να κάνετε κάποια δήλωση, σας παρακαλώ να είσαστε σύντομοι για να μην ξεπεράσουμε το χρονικό διάστημα της ε, Επιτροπής μας. Κύριε Μπρόγκς. Ακόμη και μετά από την απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου και την εφαρμογή της, νομίζω ότι ελοχεύει ακόμα ο κίνδυνος ότι η τρομοκρατία ή το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα μπορεί να συνεχίσουν να είναι ένα πρόσχημα για τη συλλογή δεδομένων. Ακόμα και όταν υπάρχει μια τέτοια υποψία για τέτοιες δραστηριότητες μπορεί τα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν για άλλους λόγους για να εφαρμοστεί παραγωγή χάρη μια απαγόρευση ουσιαστικά πολιτικών απόψεων που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη-μέλη. Η απόφαση του δικαστηρίου το εξέτασε αυτό το θέμα υπήρξε και κάτι το οποίο ελέγχθη προηγουμένως ότι η απόφαση του δικαστηρίου δεν θα ε, επηρεάσει την εθνική νομοθεσία που έχει περάσει βάσει της οδηγίας. Μήπως με τον τρόπο αυτό όμως αυτή η απόφαση του δικαστηρίου θα οδηγήσει στην εκπόνηση μιας νέας οδηγίας που θα ανατρέψει την προηγούμενη. Επανέρχομαι στον κύριο Καγιόλα. Πρώτα η Κομισιόν και η Προεδρία και μετά ο κύριος Καγιόλα για να απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα που την Η Κομισιόν πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τα διακεκριμένα μέλη για τις απόψεις που διατύπωσαν. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή χαιρέτησε την σαφήνεια που προσέδωσε ε, το δικαστήριο σε αυτή την οδηγία και επίσης σημειώσαμε ότι η απόφαση γενικά επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής του 2011 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας. Με σαφήνεια εξήγησε η νομική υπηρεσία πρωτήτερα ότι το δικαστήριο αποφάσισε ότι η φύλαξη των δεδομένων δεν ανταποκρίνεται στην αρχή της αναλογικότητας και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας. Το θέμα το οποίο έθιξε το δικαστήριο είναι πολύ σημαντικό, όπως η πρόσβαση και η χρησιμοποίηση ε, των δεδομένων από τις εθνικές αρχές, ε, επίσης ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων των πολιτών. Τα μέτρα ασφαλείας ε, για αυτά τα δεδομένα, η περίοδος και ο χώρος όπου θα διατηρούνται τα δεδομένα. Όλα αυτά τα θέματα έχουν ήδη εξεταστεί μέσα στην έκθεση αξιολόγησης τη Επιτροπής του 2011. Παράλληλα θα πρέπει να πούμε το δικαστήριο θεώρησε ότι η διαφύλαξη των δεδομένων αυτή καθεαυτή δεν επηρεάζει ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα και επίσης αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχουν σαφείς προϋποθέσεις ε, για να διαφυλάσσονται τα νόμιμα συμφέροντα και να ε, αντιμετωπίζονται περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων δημόσιας ασφάλειας και τρομοκρατίας. Ήδη η Επιτροπή έχει αρχίσει να εξετάζει την ανάγκη για μια νέα νομοθετική πρόταση και το θέμα που έθιξε το δικαστήριο είναι περίπλοκο και επίσης αυτό φάνηκε στα ερωτήματα και στην παρουσίαση που έκανε η νομική υπηρεσία. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Αυτή η εκτίμηση των επιπτώσεων θα γίνει από την Επιτροπή ε, αφού συμβουλευτεί όλους τους ε, αρμόδιες φορείς και αφού ληφθούν υπόψη όλα τα συμφέροντα τα προβλήματα που σχέση με την πιθανή αναθεώρηση ε, της οδηγίας για την, ε, την ιδιωτική ζωή και επίσης ε, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για το πλαίσιο προστασίας των δεδομένων θα ληφθούν υπόψη προτού οριστικοποιηθεί η αξιολόγηση. Γι' αυτό εμείς στην Επιτροπή προτιθέμεθα να δώσουμε χρόνο ώστε να γίνει σωστά αυτή η αξιολόγηση. Επίσης θα ήθελα να δώσω μια γρήγορη απάντηση ε, στον κύριο Ζετίνη σχετικά με τη διαδικασία παραβίασης. Θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή θα το δει ταχύτατα αυτό το πρόβλημα χωρίς καθυστέρηση και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Προεδρία, σεβόμενη τις του Δικαστηρίου, δεν έχει καθόλου σχόλια για το θέμα αυτό και σκοπεύει να συμμορφωθεί με αυτή την απόφαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καγιόλα. Δύο κουβέντε. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω η δήλωση ακυρότητα ισχύει εξ τούγκ, αναδρομικά δηλαδή, καταλαβαίνω ότι θα προκύψουν νομικέ συνέπειε από την ε, εφαρμογή τη απόφαση. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτηση τη κυρία Αρχεντίνη και του κυρίου Μωράη, Οι εθνικέ νομοθεσίε δεν επηρεάζονται αυτέ καθεαυτέ από την απόφαση. Οι εθνικοί νομοθέτε δεν έχουν πλέον την υποχρέωση να φροντίζουν για τη φύλαξη των ε, δεδομένων όπως προέβλεπε η οδηγία, αλλά μπορούν με αυτόνομες εθνικές αποφάσεις είτε να διατηρήσουν, είτε να ανακαλέσουν, είτε να ακυρώσουν οποιαδήποτε εθνικό νόμο υπάρχει σχετικά. βάσει της ακυρωμένης πλέον οδηγίας. Εάν παραμείνουν οι εθνικοί νόμοι, οι εθνικοί δικαστές θα πρέπει να αξιολογήσουν τα κατά πόσο τα θεμελιώδη δικαιώματα γίνονται σεβαστά. Άρα οι εθνικέ δικαιοδοσίε, τα εθνικά δικαστήρια τα αποφασίζουν αυτό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το μόνο που ανέλησε στην απόφαση αυτή, στην περίπτωση αυτή, με την συγκεκριμένη οδηγία, είναι ακριβώ η ίδια η οδηγία. Δεν ε, αναφέρθηκε ούτε ασχολήθηκε με άλλα νομοθετήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε σε αυτή τη φάση είναι δύσκολο να προβλέψουμε τις έμεσες συνέπειες άλλων προτάσεων ή ε, πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα για την ερώτηση της κυρίας Μπάουερ για το πώς φτάσαμε στην απόφαση αυτή πράγματι μια ένα προδικαστικό ερώτημα δύο ανώτατων δικαστηρίων που ξεκίνησαν από δικαστήριο πρωτοβάθμιο στην περίπτωση της Αυστρίας ήταν ένα λέντα της ε, Αυστριακής Ομοσπονδίας που είχε υποβάλει ουσιαστικά το προδικαστικό ερώτημα αυτά απευθύνθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπως προβλέπεται από τις συνθήκες. Έτσι, ο δικαστής, το δικαστήριο του Λουξεμβούργου μπορούσε να αποφανθεί όχι μόνο για, την, ε, το περιεχόμενο των πράξεων, αλλά και για την ισχύ τους. Πράγμα που και έγινε. Και κάτι τελευταίο που θέλω να διευκρινίσω και να επιμείνω σε αυτό το κομμάτι που μου φαίνεται αρκετά αμφιλεγόμενο. Η οδηγία που, που κηρύχθηκε άκυρη δεν είναι πλέον εφαρμοστέα. Οπότε δεν έχει νομικές συνέπειες από την στιγμή ε, θέση σε ισχύ της, ε, όπως είπα η ισχύ εξτούγκ, αλλά τίποτα δεν εμποδίζει να προταθεί νέα οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η οδηγία όμως αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμορφώνεται με τις αρχές της αναλογικότητας, οι οποίες εκτέθηκαν πολύ αναλυτικά στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο επέμεινε στην αρχή της αναλογικότητας όλος ιδιαίτερος. Ε, ανέφερε λεπτομερώ τα κριτήρια που έπρεπε να ακολουθούνται. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Προσπάθησα να συναψίσω. Ε, Εμεί σα ευχαριστούμε, κύριε Καγιόλα. Είσαστε πράγματι σύντομο. Σα ευχαριστούμε δι για αυτόν τον λόγο. Ε, να σα πω. Ήρθαμε στο τελικό τέλος αυτής της θητείας μας. Είναι η τελευταία τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Την Δευτέρα όμως στις 7 θα συνεχίσουμε με την συνεδρίαση των συντονιστών. Έχουμε ακόμη μια συνεδρίαση των συντονιστών και θα παραίσταται η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για κάποια ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν, όπως έκανα και χθες, να καταλαβαίνω την ευκαιρία στη δεξίωση που είχαμε, να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία σας, για την αφοσιωσή σας, για τη σκληρή σας δουλειά, για την ποιότητα των συζητήσεων που είχαμε και που μπορέσαμε να απολαύσουμε σε αυτά τα πέντε χρόνια που συνεργαστήκαμε μαζί ήταν μια συναρπαστική και πραγματικά ε, ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία. Και όχι μόνο για μένα. Βλέπω όμω ότι η κυρία Σαρχεντίνη θέλει ακόμα κάτι να πει πριν ευχαριστήσουμε του Γερμανεί για τα λίγα λεπτά που μα κάνουν δώρο. Όχι επειδή θέλω να έχω τον τελευταίο λόγο σε αυτή την επιτροπή μετά από τα πέντε χρόνια που διέρευσαν εσείς πρέπει να έχετε τον τελικό λόγο αλλά δεν είχα την ευκαιρία χθε, επειδή έπρεπε να φύγω βιαστικά και θα μπορέσω να το κάνω ούτε τη Δευτέρα. Θέλω όμω να σα ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο διευθύνεται τις εργασίε τη Επιτροπής μα τα τελευταία πέντε χρόνια, την υπομονή που είχατε για μας και την χαρά που μας δώσατε όταν παίξατε κιθάρα στα δίπλα μας και διασκέδασα ιδιαίτερα με τον τρόπο που μας δείξατε χθες πόσο μας εκτιμάτε. Αν ξαναγυρίσω λοιπόν σε αυτό το κοινοβούλιο, μάλλον αν δεν γυρίσω σε αυτό το κοινοβούλιο, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την δουλειά σας, την υπομονή σας, το χιούμο σας και την αφοσίωσή σας. Ευχαριστώ πολύ Γιώργη, είσαι πολύ καλή. Ούτε μπορώ να το πιστέψω. <laughs> Ελπίζω ότι θα γνωριστούμε και καλύτερα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας και καλή επιτυχία στις ε, εκλογές. Σε όλους σας που θα προσπαθήσετε να επανεκλεγείτε και καλή τύχη σε αυτούς από εσά οι οποίοι δεν θέλετε να επανεκλεγείτε και θέλω να σας δώσω ένα μήνυμα αναγνώρισης και φιλίας. Ευχαριστώ.